So, uh, uh, Συνάδελφοι, δυστυχώς ο καλεσμένος μας έχει καθυστερήσει λίγο. Ε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν ε, εξαρτιόταν από μένα θα είχαμε ξεκινήσει την ώρα μας, αλλά ο καλεσμένος μας έχει καθυστερήσει λίγο. Ωστόσο, με ενημέρωσαν ότι βρίσκεται τώρα στην είσοδο εδώ του Κοινοβουλίου, οπότε ας περιμένουμε άλλα 5-6 λεπτά. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Και δυστυχώ βέβαια ο χρόνο που έχουμε προβλέψει για αυτή τη συζήτηση είναι έω τι μισή μόνο. Δεν έχουμε όμω άλλη επιλογή. Έχετε άλλα πέντε λοιπόν ε, λεπτά στη διάθεσή σα για να καπνίσετε, να πιείτε, να μιλήσετε, οτιδήποτε θέλετε. smoke in the... Αλλά μην καπνίσετε εδώ μέσα, έτσι, στην αίθουσα.

και Okay, dear colleagues, let's start. Ας ξεκινήσουμε, συναδέλφοι. Χαίρομαι που ο κύριο ε, Πιτούκη, ο Γενικός ε, Γραμματέας της ε, ΓΕΝΚΤΑΝΤ, της Γενικής Διασκέψης των Ηνωμένων είναι εδώ μαζί μας και το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί του είναι η έκθεση εμπορίου και ανάπτυξης του 2018. Πρόκειται για μια συζήτηση που είναι κοινή μεταξύ των Επιτροπών ΔΕΒΕ και ΙΝΤΕΡ και γι' αυτό έχω εδώ εξ μου και την Αντιπρόεδρο της ε, ΔΕΒΕ, την Μύρια Καπάρεν. Ο Γενικός Γραμματέας θα μας παρουσιάσει τις, τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης με τίτλο Power Platforms and Free Trade Illusion. Νομίζω πως αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν καθημερινώς εδώ στην Επιτροπή μας, οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά το πώς το εμπόριο μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων ε, και ε, την ε, καλύτερη ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών. Οπότε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θα δώσω καταρχήν το λόγο εδώ στην Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα φινλανδικά, οπότε νομίζω πως θα χρειαστεί να βάλετε τα ακουστικά σας. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά μου κυρίσω και εγώ την έναρξη αυτής της ε, κοινή ανταλλαγής ε, απόψεων με τον ε, Γενικό Γραμματέα της UNECTAD εμείς εδώ στην, και στην δική μας Επιτροπή Ανάπτυξης εξετάζουμε συχνά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ε, ε, οι οποίες συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ε, τους επόρους τους ή να λάβουν την απαραίτητη προστιθέμενη αξία, την υπεραξία από αυτούς τους πόρους. Και ο κύριος Εκητούγη έχει αναφέρει ότι μπορεί να δοθεί υποστήριξη σε αυτές τις χώρες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως, εάν ο στόχος είναι μια τέτοια βιώσιμη ανάπτυξη η οποία συμπεριλαμβάνει τους πάντες, χωρίς δηλαδή αποκλεισμού. τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την διεξαγωγή του εμπορίου. Το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση έχουν βελτιώσει το επίπεδο εισοδήματος ε, πολλών ανθρώπων και τους έχουν ε, βγάλει από την ε, ένδια και από την άλλη, ωστόσο, πλευρά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η σχέση μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης και ένδυα αφετέρου είναι περίπλοκη. Η εξάλληψη λοιπόν της ένδυα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον εφαρμοστούν και σε εγχώριο επίπεδο οι κατάλληλε πολιτικέ. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε μια τεράστια εμ, πρόκληση. Δηλαδή πώ μπορούμε να επιτύχουμε το κατάλληλο εμπόριο χωρίς όμως να κάνουμε υποχωρήσεις, παρέχοντας δηλαδή ένα περιβάλλον το οποίο παρέχει ευκαιρίες, το οποίο περιέχει ε, δυνατότητες ε, περισσότερου ανάπτυξης για όλους. Σε ό,τι αφορά τώρα το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, το GSP, θεωρώ πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία. Πρόσφατες δηλαδή έρευνες έχουν καταδείξει ότι επιβολή μονομερών συμφωνιών GSP ε, σε ε, συνάρτηση με, τις, ε, με τους κανόνες του ΠΟΕ μπορούν να επιτύχουν πολλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει πολλά στο πλαίσιο των στόχων της και στο πλαίσιο δηλαδή του, του, του συστήματος γενικευμένου προτιμήσεων και στο πλαίσιο του συστήματος τα πάντα εκτός από όπλα, everything but arms, με αποτέλεσμα δηλαδή να μην επιβάλλεται κανένα είδους είδου δασμό στην εισαγωγή των προϊόντων από αυτέ τι χώρε. Ή εν λόγω χώρε με τη σειρά του είναι υποχρεωμένε να ε, συμμορφώνονται με τις διεθνείς συνθήκες σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, το, την προστασία του περιβάλλοντος και του ε, κανόνε χρηστή διακυβέρνηση. Θεωρώ πω ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενεργό μα συμμετοχή σε αυτό το διάλογο, ε, πάντοτε σε συνεργασία με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε το εμπόριο με βάση τις βασικές μας αξίες, τις βασικές μας αρχές. Αυτά εισαγωγικά και αναμένω με ενδιαφέρον τα όσα θα ακούσουμε σε ό,τι αφορά ε, την έκθεση της UNCTAD, σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ανάπτυξη για το 2018. Κύριε Τσούι, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η γεωγραφία δεν ήταν το φώτι μου, γι' αυτό συγγνώμη που καθυστέρησα. Με την άδειά σας δεν έχω συχνά την ευκαιρία να μιλήσω σε άτομα όπως εσάς, αλλά θα σχολιάσω και τη δουλειά μας, όχι μόνο την έκθεση. Την συνοχή μεταξύ εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής, δηλαδή τις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως ο τεχνολογικός πόλεμος όπως αποκαλείται και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Θα σας δώσω και κάποια βασικά στοιχεία βέβαια της έκθεσης. Στο κέντρο της έκθεσης μας για το 2018 βρίσκονται δύο-τρία βασικά ευρήματα. Πρώτον, η παρακολούθηση της τροτότητας ε, της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης μετά την κρίση του 2008. Εξετάσαμε και τι μορφή ανάκαμψη είχαμε. Αυτά που αποκαλούμε τα συμπτώματα της ήπιας ανάπτυξης που επιδεινώνονται από τις αυξανόμενες εντάσεις. Επίσης θα δούμε τις ε, προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας. Πρώτα-πρώτα, όπως και άλλες μελέτες έδειξαν, η αποκατάσταση της οικονομίας την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά εύθραυστη. Μετά την οικονομική κατάρρευση, κάποια θετικά αποτελέσματα απέναντι στην κρίση ήταν προϊόν πολυμερών δράσεων. Οι εντάσει, ωστόσο που διαπιστώνονται τώρα, που είναι σύμπτωμα αλλά ταυτόχρονα και πρόβλημα, μειώνουν την συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτής της εύθραυστης, όπως είπαμε, οικονομικής ανάπτυξης και προκύπτουν μια σειρά τέτοιων προκλήσεων. Στη Στην περίοδο μετά την κρίση, κάποιες βασικές αλλαγές για την ενίσχυση ενός ε, ε, προβλέψιμου καθεστώτος ανάπτυξης δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς. Τα προβλήματα της ανεπαρκούς ρυθμιστικής προσέγγισης στην περίοδο της υψηλής παγκοσμιοποίησης δεν οι αγορές ε, δεν παράγουν μόνο οικονομία αλλά και προβλήματα. Στην ουσία είχαμε μία μαζική επέκταση της παραγωγής πλούτου αλλά κακή διανομή των πλεονεκτημάτων του νέου πλούτου που παράγει το εμπόριο τόσο μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό των χωρών. Δεύτερον, και σε μεγάλο βαθμό, το εμπόριο αντιμετωπίστηκε ως ο υπεύθυνο σε μια σε έναν κόσμο με αύξηση του άγχους. Οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους για την πολιτική γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και το εμπόριο. Έχει αποδειχθεί ότι η πιο επιτυχημένη πολιτική είναι αυτή που δηλώνει ότι δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι δείγμα του ότι η παραδοσιακή μορφή πολιτικής αποτυγχάνει όταν βλέπουμε ότι η, δουλειά της πολιτικής δεν προκύπτει και άρα χρειάζεται μια άλλη μορφή πολιτικής. Ένας καλός πολιτικός λοιπόν είναι ένας πολιτικός ο οποίος δηλώνει ότι δεν θα δράσει ως πολιτικός. Ένα άλλο φαινόμενο σημαντικό στις συζητήσεις που σχετίζεται και με την αύξηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει θεσμικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει να κάνει με την ποιοτική μεταμόρφωση του διεθνούς εμπορίου. Όταν δημιουργήθηκε ο ΠΟΕ, το εμπόριο είχε αντιμετωπιστεί ως μια συναλλαγή μεταξύ χωρών παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα που πουλούν σε άλλες. Αλλά αυτό αγνοεί την απεθνικοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, διότι οι τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι πλέον η μεταφορά διαθαλάσσης κυρίως σε κοντέινερ των εμπορευμάτων ε, επέτρεψε την παραγωγή των προϊόντων πολυεθνικά από χώρα σε χώρα. Όταν λοιπόν βλέπουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών για τη διαμόρφωση των ε, συνολικών κανόνων είναι πολύ δύσκολο να πούμε τι είναι, τι γίνεται με ποια χώρα. Πάτε το iPhone. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, στον τομέα του iPhone υπάρχει διαπραγμάτευση ΙΠΑ και Κίνας για παράδειγμα, διότι η προστιθέμενη αξία του iPhone βγαίνει στην Αμερική, αλλά η παραγωγή γίνεται στην Κίνα. Άρα, η παραδοσιακή μορφή πολυμερούς διαπραγματεύσεως στα εμπορικά ζητήματα ε, αντικαθίσταται από πολλές διμερείς. Επίσης, πολλές φορές ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι η, η διαμόρφωση πολυεθνικών επιχειρήσεων με τη μορφή πολλών εθνικών εγκαταστάσεων σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πάβουν πια να έχουν μια εθνική ταυτότητα. Δηλαδή, όταν ε, ακούμε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί από τις αμερικανικές επιχειρήσεις να επαναφέρουν τις επιχειρήσεις, ε, τις δραστηριότητες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ε, έχουν φύγει από την χώρα, την αρχική χώρα προέλευσής τους, δραστηριοποιούνται παντού και επανέρχονται αγοράζοντας ε, κεφάλαιο στη χώρα προέλευσης αλλά επενδύοντας σε offshore. Αυτές είναι κάποιες από τις δυναμικές που αλλάζουν και δείχνουν ποιοι είναι, πώς εμφανίζονται οι διάφοροι δρόντες στη διεθνή οικονομία. We have Επίσης, είδαμε να αυξάνεται ο πλούτος με χωρίς να αυξάνονται τα εισοδήματα. Αυτό το αποκαλούμε συγκέντρωση πλούτου και δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο άνισων επιστροφών στις επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς μακροπρόθεσμα να αυξήσει την συσσόρευση πόλου, αλλά οι κοινωνίες κατανάλωσης δεν μπορούν να καταναλώσουν πλέον. Δηλαδή σήμερα έχουμε μικρότερη κατανάλωση, κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την μακροχρόνια βιωσιμότητα των οικονομιών. Να σας πω με δύο λόγια τις προκλήσεις που έρχονται, που έχουμε μπροστά μας. Την αύξηση της σημασία της ψηφιακής οικονομίας. Πριν όμως από αυτό, να σας δώσω και κάποια στατιστικά δεδομένα. Δημοσιεύσαμε το τελευταίο monitor της επίπτωσης των λεγόμενων εμπορικών πολέμων στην παγκόσμια κίνηση αγαθών και εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Από το 2018 μέχρι το τέλος του, το 17 μέχρι το του τα πρώτα στατιστικά δεδομένα δείχνουν δύο τάσεις. Πρώτον, το παγκόσμιο εμπόριο είναι το πιο εξαγωγικό εμπόριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. 19,63 δολάρια. Αυτή η αύξηση των εξαγωγών πώς εξηγείται από τη συνύπαρξη άγχους και προβληματισμών για το εμπόριο. Η απάντηση είναι ότι η οι επιχειρήσεις των ΙΠΑ αύξησαν κατά 40% τις εξαγωγές του προς, προς τις ΙΠΑ εν αναμονή ή προβλέποντας τον εμπορικό πόλεμο με τις ΙΠΑ. Διότι προφανώς ε, είναι διαφορετικό να χρειαστεί να, πληράσει, να πληρώσεις δασμούς 10-20% ανάλογα με το πότε θα στείλεις τα προϊόντα σου στις ΗΠΑ Βέβαια, αυτοί που χάνουν από τους εμπορικούς πολέμους ήταν οι χώρες του ΑΣΕΑΝ, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία. Και ποιος είναι ο λόγος. Είναι μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών που έχουν την αλυσίδα παραγωγής τους μέσω Κίνας. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται άμεσα και απευθείας, ιδίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, από την ε, επαναφορά των, από την αλλαγή των δικτύων παραγωγής ε, ανάλογα με τις ε, αυξομοιώσεις των δασμών. Η δεύτερη κατηγορία αυτών που χάνουν είναι η ΙΠΑ και η Κίνα. Και αυτοί που κερδίζουν είναι οι Ευρωπαίοι. Πρώτα, η Βραζιλία και η Ινδία κατόπιν. Και αυτό είναι κατανοητό. Τα προϊόντα που θέλει να εισάγει η Κίνα από τις Πολιτείες και δεν μπορεί να τα εισάγει πλέον από εκεί, τα εισάγει από την Ευρώπη. Και, και στην Ευρώπη όταν εισάγουν από την Κίνα ή δεν μπορούν, όταν δεν μπορούν πια να εισάγουν από την Κίνα, τα εισάγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα οι, αυτοί που, που κερδίζουν είναι οι Ευρωπαίοι, Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία. Τώρα, η συγκέντρωση αν μας ανησυχεί η συγκέντρωση της ε, κυριαρχίας σε κάποιες εταιρείε που αποκτούν ε, ηγεμονικό χαρακτήρα στο παγκόσμιο εμπόλιο, αυτό έχει επιπτώσεις και στην ψηφιακή οικονομία. Διότι υπάρξει ταχεία αύξηση των πλατφορμών ε, ψηφιακής ε, οικονομίας που αντικαθιστούν πολύ γρήγορα τους παραδοσιακούς γίγαντες του εμπορίου και δεύτερον λόγω της μαζικής συγκέντρωσης ε, πλούτου και δυσανάλογης επέκτασης του πλούτου σε σχέση με την αύξηση της εργατικής, του εργατικού δυναμικού. Τι βλέπουμε λοιπόν. Διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης. Π.χ. οι μεγαλύτερες 25 πολυεθνικές σήμερα είναι κατά βάση ε, ψηφιακού χαρακτήρα. 14 Αμερικέ, 3 ευρωπαϊκέ, 3 Κινέζικες, μία από την Αφρική, μία από την υπόλοιπη Ασία. Αλλά και εκεί ο μέσο πλούτο είναι 400 δι για τι αμερικανικέ, 200 δι για τι ε, Κινέζικες, 1,3 δις για την, άλλη Κινέζη, για την άλλη Ασιατική και πολύ λιγότερα για την Ευρώπη και την Αφρική. Και τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, το μέλλον είναι στο, στην ψηφιοποίηση. Αλλά αποφεύγοντας τα λάθη που κάναμε στην παγκοσμιοποίηση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυνατότητες καλύτερων αποδόσεων και πιο δίκαιων αποδόσεων του κέρδους των, της ψηφιακής, του, του ψηφιακού εμπορίου, της ψηφιακής δραστηριότητας στην οικονομία. Αν αρχίσουμε απλά και λέμε ότι η ψηφιακή οικονομία είναι κακή και δεν αντιμετωπίσουμε την ψηφιακή, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αναπτυσσόμενων και ε, αναπτυγμένων οικονομιών, θα έχουμε κάνει τεράστιο λάθος. Το λέω αυτό γνωρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν έδειξε μόνο παγκόσμια ηγεσία στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει την, ε, τις ανισότητες της ψηφιακής οικονομίας, αλλά είναι και πρωτοπόρο στην ε, διευκόλυνση των ε, ε διασυνοριακών μεταβιβάσεων στην ψηφιακή, οικονομία. Εμείς είμαστε υπέρ της... Εσείς είσαστε υπέρ της προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης της ψηφιακής δραστηριότητας. Και αυτά θα είναι στο κέντρο της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να είναι και μπροστά στην ψηφιακή οικονομία και μπροστά στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Έχουμε λίγο χρόνο τώρα στη διάθεσή μας για να διεξάγουμε συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας, η Μαρία Ρενά πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πρέπει να πω ότι είμαι θειασότης, υπέρμαχος όλων αυτών των εκθέσεων που έχουμε από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, διότι οι εκθέσεις αυτές μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για εμάς τους πολιτικούς. Πληροφορίες που πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε λίγο περισσότερο την πολιτική που ακολουθούμε. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το εμπόριο όντως μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την υποστήριξη της ανάπτυξης, αρκεί το εμπόριο να διεξάγεται μέσω μιας μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμης πολιτικής και οράματο και να μην προσεγγίσουμε το εμπόριο μόνο βραχυπρόθεσμα, δηλαδή με απόλυτο στόχο μόνο το να πλουτίσουν ορισμένοι και να δημιουργηθούν συστηματικά κέρδη για συγκεκριμένα μονοτμήματα του πληθυσμού και δυστυχώ ακριβώ αυτό βλέπουμε σήμερα. Και στην ίδια την έκθεση λέγεται ότι το εμπόριο όπως ε, υλοποιείται αυτή τη στιγμή με το εμπορικό μοντέλο το οποίο ακολουθούμε αυτή τη στιγμή παγκοσμίω, ουσιαστικά ενισχύει την όλη ιδέα της ε, απόδοσης της κερδοφόρας σε συγκεκριμένες μόνο πολυεθνικές ενισχύει το εμπόριο, το σύστημα αυτό μέσω της ε, κερδοφορίας όπως αυτή διαμορφώνεται στις χρηματοπιστωτικές ανταλλαγές αλλά και στην πνευματική διοκτησία το είπατε και εσείς αυτό πριν από λίγο. Το εμπόριο όπως υλοποιείται αυτή τη στιγμή ενισχύει όλα αυτά τα συστήματα DSCS ή ICS για τη συγκεκριμένη προστασία συγκεκριμένων επενδυτών και επίσης το εμπόριο με την φυστάμενη μορφή του ουσιαστικά συμβάλλει στο να έχουμε πολύ έντονες ανισότητες παγκοσμίως. Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν στρέφομαι κατά του εμπορίου, αλλά κατά του υφιστάμενου εμπορίου, του εμπορίου που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρώ ότι είναι Ευαγγέλιο για μένα οι εκθέσεις της UNCTAD όσον αφορά την προτινόμενη εμπορική και επενδυτική πολιτική και ανέκαθεν τις ακολουθούσα στο πλαίσιο της εντολής μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την υπερπαγκοσμιοποίηση στην οποία αναφερθήκατε, το ότι έχουμε μια φοβερή αύξηση των πολυεθνικών εταιριών και της παρουσίας τους στην παγκόσμια οικονομία, ακριβώς για αυτό το λόγο θέλαμε εμείς να εντάξουμε περισσότερο στην παγκόσμια οικονομία και τις εμπορικές συμφωνίες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θελήσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή ένα κεφάλαιο που να λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικά πρότυπα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, διότι αν πραγματικά θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Και για ακόμη μια φορά έκθεσε αυτή λέξη ξεκάθαρα το εμπόριο, με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή, μολονότι μπορεί να έχει οδηγήσει σε κέρδη σε ορισμένα μέρη του κόσμου, από την άλλη πλευρά είναι υπέτειο για τη δημιουργία ανισοτήτων ή για την ενίσχυση των ήδη φυστάμενων ανισοτήτων και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην Ευρώπη οι κοινοί γνώμη, οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια ή σκεπτικισμό τις εμπορικές αυτές συμφωνίες ακριβώς επειδή θεωρούν ότι έχουν παραγωνιστεί από τις συμφωνίες αυτές, ότι έχουν μείνει εκτός. Όσον αφορά το κέρδος, πάρα πολλοί λένε ότι τα κράτη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να το κατανείμουν ισότιμα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο μέρος του κέρδους το οποίο διαφεύγει από το ίδιο το κράτος μέσω της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Άρα το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να κατανείμει προφανώς τον πλούτο που του διαφεύγει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εμπορικές αυτές συμφωνίες ως εργαλεία τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν, θα πρέπει να εμπεριέχουν συγκεκριμένε ρήτρε κατά τη φοροδιαφυγή, θα πρέπει να εμπεριέχουν ρήτρε που να προβλέπουν ότι θα τηρούνται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και εν τέλει αυτό το οποίο λέμε εδώ και τέσσερα χρόνια στην Επιτροπή αυτή είναι ότι δυστυχώς ε, οι φιλελεύθεροι συναδελφοί μας και οι συντηρητικοί συναδελφοί μας δεν ακούνε καθόλου τις απόψεις αυτές. Κύριος, κυρία Χόιμπακ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση που μας κάνατε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφος Μαρία Αρένα. Συμφωνώ δηλαδή πλήρω με την ανάλυση που κάνατε και μπορούμε πάντοτε να βασιζόμαστε στι εκθέσει σα όταν συζητούμε την αναπτυξιακή πολιτική. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή η ψηφιοποίηση. Ε, το, το ε, ζήτημα βέβαια εδώ σε σχέση με την ψηφιοποίηση ε, είναι το πού ακριβώς βρίσκονται τα σχετικά δεδομένα, συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα μέρη του κόσμου ή θα πρέπει να είναι πιο αποκεντρωμένα τα δεδομένα και να απαντούνται σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Εάν θέλουμε τα δεδομένα αυτά να βρίσκονται στην κατοχή και στην κυριότητα εκείνων στους οποίους ανήκουν αυτά τα δεδομένα, ε, τότε θα ήθελα να μου πείτε ε, ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά στις διαδραματεύσεις που γίνονται αυτήν την περίοδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου. Επίσης, τι συμβαίνει στο πλαίσιο, για παράδειγμα, διαδικασιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν χώρε στι οποίε το δημοκρατικό πολιτεύμα δεν λειτουργεί καλά, με αποτέλεσμα τα δεδομένα αυτά να αξιοποιούνται όχι μόνο για να προωθείται η περιφερειακή οικονομία, αλλά και προκειμένου να ασκούνται πιέσει στου πολίτε. Και προκειμένου να γίνεται κατασκοπία, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, ει βάρο των πολιτών. Άρα λοιπόν ένα ακόμα ερώτημα που τίθεται είναι ε, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε από τη μία πλευρά την ελευθερία στο διαδίκτυο, αλλά από την άλλη πλευρά να μην αξιοποιείται το διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση ει βάρο των πολιτών. Και ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξή. Αναφερθήκατε στην ανισορροπία, αν θέλετε. Ανισορροπία ουσιαστικά δηλαδή αφορά τη Δύση αφενός και τη λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αφετέρου. Μια ανισορροπία την οποία αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ. Ε, στην Δύση. Οπότε, ε, ποια θεωρείτε ε, πως θα πρέπει να είναι η υποχρέωση που θα βαρύνει σε ό,τι αφορά με τη σχετική ε, τις επιχειρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ελεύθερες, ελεύθερα συναπτώμενες συμβάσεις σε ό,τι αφορά για παράδειγμα διατάξεις που αφαιρούν το περιβάλλον, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής ή θα πρέπει να υπάρχει κάτι πιο δεσμευτικό. Και αυτό ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό κόσμο θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σα άποψη. Αυτά και σα ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος ο κύριο Σόλτ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ από την πλευρά μου να σας καλωσορίσω θερμά. Εμείς κατά την τελευταία σύνοδο της ε, διάσκεψης στον Αερόμπι, είχαμε τη δυνατότητα να περιβρεθούμε και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο-τρία ζητήματα. Σε ό,τι αφορά ε, την ανάγκη αντιμετώπισης νέων ε, ρυθμιστικών προκλήσεων σε σχέση με τις ψηφιακές ειδικότερα πλατφόρμες, να πω ότι σε ό,τι αφορά ορισμένες επιχειρήσεις υπάρχει και μια συμπεριφορά από την πλευρά αυτών των επιχειρήσεων η οποία υπονομεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και αυτό μας οδηγεί στο ε, ερώτημα, αν θέλετε, στο ζήτημα των κινήτρων τα οποία υποτείνουν αυτή τη συμπεριφορά από τον, αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή την διατήρηση και τη μεγέθυνση του μεριδίου της αγοράς τους. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τα παγκόσμια οικονομικά συστήματα καθίστανται πιο ευάλωτα, πιο ευπαθή και αυτό που σας ρωτάω είναι πώς θεωρείτε με βάση το σημερινό οικονομικό σύστημα, παγκόσμιο ε, οικονομικό σύστημα, πώς θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, ρυθμιστικές ε, προκλήσεις και πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία για, τον, για την εποχή, αν θέλετε, της ψηφιοποίησης. Δεν θα πρέπει δηλαδή να ενισχύσουμε την ικανότητά μας σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της δραστηριότητας την οποία ασκούν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεύτερο ερώτημα. Ε, στην έκθεσή σας αναφέρεστε ε, στην αντιμετώπιση των ασυμμετριών που υφίστανται σήμερα στις αγορές. και την ε, δημιουργία Ε, και ψηφιακών πλατφορμών οι οποίε βρίσκονται στις, στις, σπάγαν ακόμα στι απαρχέ τη δημιουργήση του. Εδώ έχουμε την αντιμετώπιση από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων τέτοιων νέων ψηφιακών πλατφορμών ή ως δημοσίων ε, πλατφορμών ή ως ε, πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οπότε έχουν, έχουν, θεωρείται πως έχουν υπάρξει κάποιες απόπειρες μέχρι στιγμής για να αντιμετωπιστεί αυτό το ε, φαινόμενο. Δηλαδή θεωρείται πως κυβερνητικές επανεμβάσεις στον τομέα του, τον ψηφιακό είναι δικαιολογημένε ακριβώς για να ε, αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, συγκέντρωση δύναμης από την πλευρά ορισμένων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. το λόγο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Ε, και νομίζω πως ε, ήδη αναφέρθηκε αυτό, ότι δηλαδή ε, ναι μεν θέλουμε εμπόριο για όλου, αλλά η ευημερία τελικά που προέρχεται από το εμπόριο δεν αποβαίνει προ όφελο ε, όλων και όπω ήδη αναφέρθηκε από άλλου συναδέλφου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτέ τι πρακτικέ. θα πρέπει να ε, βρούμε βιώσιμε λύσει. και αν δούμε ε, τις ε, συμφωνίες τις οποίες συνάψαμε πρόσφατα από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τότε διαπιστώνω ότι δεν ακολουθούμε την κατάλληλη άγουσα δηλαδή ε, περιλαμβάνουμε μεν ένα κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη, αρχίζουμε να αναφερόμαστε σε ζητήματα καταπολέμηση τη διαφθορά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότιμη μεταχείριση των φύλων, καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και ε, προστασία του περιβάλλοντο και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Αλλά όλε αυτέ οι συμφωνίε ε, βασίζονται σε προαιρετικές ρυθμίσεις και βασιζόμαστε, αν θέλετε, στην εκτίμηση ότι η εταίρος μας θα εφαρμόσει με τον ίδιο τρόπο αυτές τις διατάξεις με αυτό που τον εφαρμόζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι προς εσάς, θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις. Μήπως δηλαδή θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το εμπόριο έτσι ώστε να επιτύχουμε πραγματικές αλλαγές στις χώρες με τις οποίες έχουμε τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Και νομίζω πω ε, αυτό που αναφέρθηκε μόλι τώρα είναι πολύ σωστό ότι δηλαδή συχνά διαπιστώνουμε ότι οι μεγάλε επιχειρήσει είναι εκείνε οι οποίε επωφελούνται από τέτοιου είδου συμφωνίε. Πώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτέ τι διαδικασίε και τι μικρέ επιχειρήσει. Η ψηφιοποίηση δηλαδή προχωράει όλο και περισσότερο. Οπότε ε, θέλαμε να ακούσουμε ποιε είναι οι δικέ σα προτάσει ω προ αυτό. Δηλαδή πώ στο πλαίσιο τη ψηφιοποίηση θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα ωφέλη και για τι μικρότερου, για του επιχειρήσει και όχι μόνο για τι πολύ μεγάλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα της UNCTAD για την έκθεσή του που δίνει πραγματικά φρέσκες ιδέες για το ζήτημα. Και εδώ ίσως είναι σημαντικό να δούμε τις διαφορές δράσεις της UNCTAD και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η UNCTAD καλύπτει όλο τον κόσμο και δεν ασχολείται μόνο με το εμπόριο αλλά και με την ανάπτυξη. Όπως βλέπουμε και από την έκθεση, πέραν των πολυεθνικών ε, η έκθεση της UNCTAD μιλά για τους πολίτες και ελπίζω οι συνάδελφοι να ακούσουν το μήνυμα που ήρθε από τον Γενικό Γραμματέα της UNCTAD. Στον ψηφιακό κόσμο αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι κανόνες είναι πολύ λίγοι. Αυτό ενισχύει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εις βάρος των κρατών. Έχω τώρα μια σειρά ερωτήσεων. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το πλέγμα νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων ώστε να προστατεύσει τους πολίτες από την, ε, τις καταχρήσεις του ψηφιακού κόσμου. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα επίπεδο ισότιμης μεταχείρισης σε όλο τον κόσμο. Πώς θα το πετύχουμε αυτό στην Κίνα η εκμετάλλευση των δεδομένων είναι πολύ λιγότερο περιορισμένη από ό,τι στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές για να διαμορφώσουν ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να προστατευθούν και να αναπτυχθούν στον ψηφιακό κόσμο. Μια τελευταία παρατήρηση. Μήπως ο ΙΕ ή η UNCTAD θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στον τομέα, το, στον αυτό και θα σας άρεσε μια τέτοια ιδέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Κιτούγη για την παρουσία του εδώ. Ο τίτλος της έκθεσης το, τα λέει όλα. Η εξουσία των πλατφορμών και η χήμερα του ελεύθερου εμπορίου. Εγώ θα περίμενα μόνο από τον τίτλο να σηκωθούν να φύγουν. Δεν θέλουν πολιτικές ομάδες να συζητήσουν κάτι τέτοιο πόσο μάλλον να τα λύσουν. Δύο ερωτήσεις. Στη σελίδα 96 της έκθεσης αναφέρεται ότι οι χώρες πρέπει να προχωρήσουν πολύ προσεκτικά όταν υπογράφουν συμβάσεις για ψηφιακή οικονομία ή δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου γιατί δεν γίνονται κατανοητές οι επιπτώσεις τέτοιων τεχνολογιών στο μέλλον. Ενδεχομένως δηλαδή κάποιες χώρες που υπογράψουν κάτι τέτοιο σήμερα να το μετανιώσουν αργότερο. Εμείς είδαμε τις επιπτώσεις που είχε η υπογραφή της συμφωνίας του Μαρακές ε, και η ερώτησή μου έχει αυτή η προειδοποίηση στη ΣΟΚΤΑΤ τι συνέπειες έχει στην όψη της προσεχούς ε, μεταρρύθμισης του ΠΟΕ. Δεύτερον, διαβάζω φράσεις από την έκθεση. Το ελεύθερο εμπόριο απέδειξε να είναι ένα ιδεολογικό φύλλο πορείας που άφησε που αγνόησε τις πολιτικές, την πολιτική βούληση των αναπτυσσομένων χωρών και μείωσε τις, ε, τα εισοδήματα των χωρών αυτών. Αυτό συμβαίνει, το ξέρουμε. Προτείνεται ωστόσο τρεις προτεραιότητες δράσης σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. Σύνδεση των διαπραγματεύσεων με δέσμευση πλήρους απασχόλησης και αύξηση ε, μισθών, ε, αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των μεγάλων επιχειρήσεων και επαρκές πολιτικό πλαίσιο ούτως ώστε οι, ανεπιξα... οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να διαχειριστούν τον πολιτικό τους χώρο. Εσάς λοιπόν, εσείς Γενικός Γραμματέας της UNCTAD, τι άποψη έχετε περί αυτού? Τι άποψη έχετε για τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ένωση, ιδίως στο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας. Σήμερα το πρωί εδώ εγκρίναμε την αναβίωση της εμπορικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, το TTIP. Φαίνεται ότι ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Η ερώτησή μου είναι, πιστεύετε ότι το μοντέλο συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου που προωθεί η Ένωση οδηγεί σε μεγαλύτερη καταστροφή σε ανισότητες. Τι μας συμβουλεύετε να κάνουμε αντί για αυτές. Ευχαριστώ. Κύριο Ζουρουμπίχ. Äh, Σας ευχαριστώ θερμά. Θα συμφωνήσω μετά όσα είπε η συνάδελφο δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να προωθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ιδιαίτερα οι οικογενειακέ επιχειρήσει παίζουν εδώ σημαντικό ε, ρόλο και συνήθω σε αυτέ τι οικογενειακέ επιχειρήσει οι γυναίκε είναι εκείνε οι οποίε διασφαλίζουν ε, την ευημερία ε, της ε, οικογένειας. Πάντοτε βέβαια αυτό το ζήτημα έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά δηλαδή γνωρίζουμε πως όταν ε, παράγουμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε και μπορούμε να τα πολλούμε, αυξάνουμε την ευημερία μας και την αγοραστική μας δύναμη. Από την άλλη όμως πλευρά ε, ισχύει και το ότι οι οικογένειες θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές για τις αγορές τους. Γιατί όσο φτηνότερα αγοράζουν, τόσο υψηλότερη αγοραστική δύναμη έχουν. Άρα λοιπόν, έχουμε από τη μία πλευρά τις την, την, την, ε, τις ε, φτηνότερες και από την άλλη πλευρά τις εξαγωγές του πλεονάσματος που οδηγούν τελικά σε διπλασιασμό της ε, ε αγοραστικής δύναμης. Και ακριβώς αυτό το Aid for Trade στο πλαίσιο και του ΕΠΟΕ σε αυτό στοχεύει. Στην υποστήριξη δηλαδή των εργαζομένων έτσι ώστε και με περαιτέρω κατάρτιση και με περαιτέρω γνώσεις να μπορούν να παρέχουν να παράγουν περισσότερα προϊόντα τα οποία θα πολλούνται και εκτός της χώρας τους. Ε, Εμένα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στόχο ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα η βιώσιμη ε, παραγωγή τροφίμων, ε, δηλαδή στη γεωργία. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ε, παραγωγή τροφίμων σε βάθος χρόνου επίσης. σε ό,τι αφορά τον στόχο 6, την, την, διασφάλιση των απαραίτητων υδάτων, τον, τον καθαρισμό των λιμάτων, και ε, το ζήτημα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρείτε πως ε, μπορούμε μέσα στο νέο, στα νέα προγράμματα να θέσουμε προτεραιότητα σε όλα αφορά τις επενδύσεις, ειδικότερα σε υπαίθριες περιοχές, σε αγροτικές σε περιοχές, όπου θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο οι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, θα είμαι σύντομο. Καταρχήν σα ευχαριστώ πολύ για τα όσα μα παρουσιάσατε. Ε, ε, στο τέλο τη παρέμβασή σα, ταχθήκατε υπέρ ενό νέου πολυμερού συστήματο ε, θεωρείται όμως υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη από την πλευρά όλων, γιατί αυτό που παρατηρούμε τη σήμερα ημέρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ σημαντική και έντονη ε, εμπορική διαμάχη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, δύο πολύ μεγάλους ε, παίκτες. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται μεν στην, στο πολυμερέ εμπόλιο, το πολυμερέ σύστημα, αλλά ουσιαστικά στην πράξη συνάπτει συμφωνίε οι οποίε απέχουν πολύ από αυτήν την πολυμερή προσέγγιση. Αναφερθήκατε και στι ε, αναπτυσσόμενε χώρε, οι οποίε συχνά δεν αναλαμβάνουν το ρόλο που θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτή τη προσπάθεια. Οπότε, ε, πού θεωρείτε πω πρέπει να γίνουν κάποιε προσπάθειε για να επιτύχουμε αυτό το πολυμερέ σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαντλέν. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καθηγητά κύριε Κιτούγη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα σήμερα. Να αντιδράσω λίγο σύντομα στα όσα λέγονται στην έκθεση αυτή. Δεν θα σας προξενήσουν εντύπωση τα όσα θα πω, γιατί τα είπα άλλωστε και στη Γενέβη. Καταρχάς, να πούμε ότι ευχαριστούμε την UNCTAD για όλη την εμπειρογνωμοσύνη που έχει δείξει στον τομέα του εμπορίου και της ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά το ρόλο του εμπορίου και των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αναφέρεστε εδώ πέρα εσεί ιδίω στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε που μπορούν να αποφεληθούν από το εμπόριο. Σε σχέση όμω με την έκθεση αυτή, θα θέλαμε να εκφράσουμε τι ανησυχίε που είχαμε εκφράσει και στη Γενέβη τον Οκτώβριο, αλλά και πρόσφατα στην εκτελεστική συνεδρίαση του, α, της Επιτροπής Ανάπτυξης. Λυπούμεθα για τον ιδιαίτερα επικριτικό τόνο που είχε έκθεση αυτή, καθώς επίσης και για το ότι με ιδιαίτερη ελευθερία αποσαφηνήθηκε η, η ευρύτητα, αν θέλετε, της έκθεσης αυτής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ξεκινάτε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καλύπτεται τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 80 και το καθεξής. Επίσης έχουμε κάποιες συγκεκριμένε παρατηρήσεις όσον αφορά τα ευρήματα, τα πορίσματα της έκθεσης αυτής, ιδίως όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης γίνονται πολλές επικριτικές αναφορές όσον αφορά την εργασία που γίνονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου όσον αφορά τα ψηφιακά ζητήματα, εμείς θεωρούμε ότι υπερβαίνεται εδώ πέρα την εντολή της UNCTAD, καθότι αναφέρεστε σε αποφάσεις που λαμβάνουν κυρίαρχα κράτη στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επίση, δεν είναι αρκετά ισορροπημένη, θεωρούμε, η εκθεσή σα. Σε κάποια σημεία αναφέρεστε σε κάποιε αφηρημένε απειλέ, ενώ σε άλλα σημεία δίνετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώ η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να χειραφετήσει πραγματικά του πολίτε. Επίση, απουσιάζουν κάποιε πιο επικοδομητικέ πληροφορίε. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια έκθεση της UNCTAD, η οποία ουσιαστικά μεροληπτεί από ιδεολογικής πλευράς και θα έλεγα ότι ακόμα και στη διατύπωσή της, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, είναι αρκετά προκλητική. Νομίζουμε ότι αυτό δεν προωθεί τον ρόλο που θα πρέπει να έχει η UNCTAD, η οποία θα πρέπει να ήταν μια διάσκεψη ουσιαστικά αμερόληπτη, αντικειμενική, η οποία να συμβάλλει πραγματικά στην όλη συζήτηση που γίνεται για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Νομίζω επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα ανάμεσα στην έκθεση αυτή καθεαυτή και την σφαιρική ανασκόπηση που γίνεται επίση από την Γενική Διάσκεψη για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη. Βλέπω ότι δεν σας προκαλούν εντύπωση τα όσα λέω αυτή τη στιγμή γιατί τα έχω επαναλάβει και σε προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας thank you very much. Uh, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το τελευταίο σχόλιο που κάνατε. Όντως, ε, καταγράφω τα όσα είπατε και βέβαια ανάλογη ήταν και τη δρασή μου την πρώτη φορά που ε, μου είπατε τα όσα μου είπατε. Θα έλεγα ότι στον οργανισμό μας έχουμε συγκεκριμένα τμήματα και 10 ετήσιες εκθέσεις, δημοσιεύσεις θα έλεγα ότι μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις είναι αυτές, αυτές που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό κόσμο, την ψηφιακή οικονομία, την οποία δημοσιεύουμε εδώ και αρκετά χρόνια και παρακολουθούμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται, αν θέλει, το ψηφιακό οικονομικό κόσμο. Θα έλεγα ότι είμαστε ο βασικό οργανισμό στα πλαίσια των ΗΕ που προσπαθούν να βοηθήσουν να αναπτυσσόμενε χώρε να γεφυρώσουν το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. Και μην ξεχνάμε ότι ε, γίνονται διάφορες μελέτες που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή ετοιμότητα των αναπτυσσομένων και των λιγότερων αναπτυγμένων κρατών. Και ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ποιε είναι οι λήψει των κρατών αυτών, ε, ποιε είναι οι απαιτήσει που υπάρχουν σε δεξιότητε προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν και αυτέ ψηφιακά, τι συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, με, τα, με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ε, χώρες στα ζητήματα αυτά. Τώρα η έκθεση που έχει να κάνει με το εμπόριο και την ανάπτυξη ουσιαστικά είναι μια μακροοικονομική επισκόπηση του πώς έχουν τα πράγματα. Δεν κάνουμε προτάσεις και συστάσεις πολιτικής για το μέλλον στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Και έτσι λοιπόν, ενώ ορισμένοι στην έκθεση αυτή βλέπουν ε, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες αρνητικές εκτιμήσεις εμείς δεν στρεφόμαστε προφανώ κατά τη ψηφιακή οικονομία. Αντίθετα, θα μπορούσα να σας πω ότι προωθούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο φορέα το ζήτημα της ψηφιακής οικονομίας και της ισότιμη χρησιμοποίησης των πόρων στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας. Αυτή ήταν η στάση που ανέκαθεν ακολουθούσαμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το είπατε, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στα όσα λέμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, διότι υπερβαίνουμε ενδεχομένω την εντολή μα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Είμαστε και εμεί ισότιμο μέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και μην ξεχνάμε ότι στα πλαίσια τη UNCTAD εκπαιδεύουμε και διαπραγματευτέ στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για ζητήματα όπω το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ουσιαστικά του λέμε ότι αν ασχοληθούμε με το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να εστιαστούν στα εξή ζητήματα. Ότι υπάρχουν τα εξή κακό κείμενα, κείμενα τα οποία θα πρέπει να θεραπευθούν και ότι θα πρέπει να προωθήσουν συγκεκριμένε πολιτικέ μέσω των οικονομικών πολιτικών. Του εξηγούμε επίση ποιοι είναι οι βασικοί του συνομιλητέ, αν θα πρέπει να ασχοληθούν κυρίω με τι ψηφιακέ πλατφόρμε, μήπω θα πρέπει να κοιτάξουν και λίγο πιο πέρα από τι κυβερνήσει, να δούνε και άλλου συνομιλητέ πέρα από του κρατικού αξιωματούχου. Ακριβώ αυτό προσπαθούμε εμεί να κάνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλου αυτού του διαπραγματευτέ στον τομέα των διαπραγματεύσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καταρχάς, ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Σας ευχαριστούμε για τις ε, παρεμβάσεις σας, τις θετικές σας δηλώσεις. Εντάχει να φερθώ σε κάποια ζητήματα. Γίνεται πάρα πολλής λόγος για την μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Εμπορικού Συστήματος. Προφανώς χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Αλλά αν έχουμε διαφορετικέ χώρε και διαφορετικού συνομιλητέ που προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, ε, τότε δεν πάμε πουθενά. Ορισμένα αναφέρονται σε ζητήματα που άπτονται του 21ου αιώνα, όπω το ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλοι θέλουν μεταρρυθμίσει προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα στα πλαίσια του κύκλου διαπραγματεύσεων τη Δόχα. Άλλοι λένε ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ προκειμένου να προστατευτούν και να προωθηθούν περισσότερο τα πνευματικά δικαιώματα και όχι τόσο πολύ οι δασμοί για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Πολλέ διαφορετικέ μεταρρυθμίσει θέλουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η σημαντικότερη πάντω πρόκληση νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι οι περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να περασπιστούν πλέον τις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις. Μιλάνε για πολυμερές σύστημα, αλλά στην πράξη δεν προωθούν το σύστημα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο των καιρών και καταδεικνύει τελικά ότι δεν υπάρχει πλέον επαρκής εμπιστοσύνη στο πολυμερές εμπορικό σύστημα. Εμείς μέσω της UNCTAD προσπαθούμε να δείξουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίζεται μόνο σήμερα λέμε ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε συγκεκριμένες αδυναμίες που έχουν να κάνουν με το σύστημα μεταρρυθμίσεων, οι οποίες όμως αδυναμίες εμφανίστηκαν και πριν από 50 χρόνια. Αυτό λέμε και στην έκθεση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ουσιαστικά βασίζεται και στην συνθήκη της Αβάνας όπου προβλεπόταν εκεί πέρα ένα ισότιμο σύστημα προστασίας των ε, κρατών στα πλαίσια του παγκόσμιου εμπορίου. Τέτοιες προσπάθειες λοιπόν διεθνείς έχουν γίνει και στο παρελθόν. Και στο παρελθόν πριν από 50 χρόνια πιστεύαν ορισμένοι θα μπορούσαμε να πειθαρχήσουμε, αν θέλετε, το παγκόσμιο εμπορίο προκειμένου να λειτουργεί υπέρ όλων με τρόπο ισότιμο. Και αυτό το οποίο λέμε στην έκθεση είναι ότι η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε τελικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από το παρελθόν. Και κάτι ακόμα. Αληθεύει ότι όντω υπάρχουν σημαντικέ προκλήσει όσον αφορά τα βιομετρικά στοιχεία, τα big data, το ζήτημα τη προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Και όντω υπάρχουν επιχειρήσει που μπορούν να καταχραστούν τελικά όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν για του πολίτε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι κυβερνήσει. Λέμε ότι θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Κάτι ακόμα. Οι παρεμβάσει των κυβερνήσεων, ξέρετε ότι παρουσιάζουν και αυτέ διακυμάνσει με, το πόσο, με βάση το πόσο ισχυρέ είναι οι κυβερνήσει. Τι τελευταίε εβδομάδε είδαμε κάποια απτά παραδείγματα. Σα ζητώ συγγνώμη, έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ, λέει η Συμπρόεδρο. Πολύ ωραία. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου απλώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Άκουσα τόσο τι επικρίσει σα όσο και τα θετικά σα σχόλια. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προσπαθώντα να στείλουμε ένα λογικό ηχηρό μήνυμα και κυρίω ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να είναι συλλογικό, να εκπροσωπεί όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Ευχαριστούμε. Ε, ε, και τον προσκεκλημένο μας και τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές παρασυμβάσεις τους και τις ιδιαίτερα ε, απαιτητικές ερωτήσεις που θέσατε και τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Κλείνουμε αυτό το τμήμα της ε, συνάντησης. Να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός διεθνούς βιώσιμη, ε, βοήθειας, αλλά αυτό πρέπει να είναι προς όφελος και των αναπτυσσόμενων χωρών και με στόχο να βοηθήσουν το εμπόριο και την ανάπτυξη. Ο κύριος Κουτικητούργη υπογράμμισε ιδιαίτερα την σημασία της ψηφιακής οικονομίας. Είμαι βέβαιος ότι μας έδωσε τροφή για σκέψη στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους σας και τον κύριο Κιτούη ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια.